Die Επαναρχίζουμε τη συνεδρίασή μα. Υπάρχουν αντιρρήσει στην ημερήσια διάταξη. Εάν όχι, έχουμε εγκρίνει τα πρακτικά. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο τη ημερήσιας διάταξη, που είναι η συζήτηση.